Ε, Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την τρομερή μου καθυστέρηση αλλά βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι έπεσαν στο ίδιο πρόβλημα που είχα και εγώ, δηλαδή τη διαδήλωση που βλοκάρισε όλη την ε, πόλη. Για την ημερήσια διάταξη πρέπει να σας πω ότι ο συνάδελφος Λίζεκ έχει σοβαρά, σοβαρά προβλήματα και πρέπει να φύγει. Το σημείο λοιπόν του κυρίου Λίζεκ θα συζητηθεί στο σημείο 4 αντί του σημείου 8 για να μπορέσει να φύγει. Θα συζητήσουμε δηλαδή αμέσως ε, μετά την εξέταση της ε, έκθεσης ε, σχετικά με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ισλανδία. Για την χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της 4ης και 5ης Δεκάτου. Και αν δεν έχετε προβλήματα, δεν έχετε ερωτήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, ούτως τροποποιημένη. Τώρα, μοιράστηκε σε όλους ε, το χρονοδιάγραμμα του 2012, σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας και να ε, κρατήσετε, να κλείσετε τις ημερομηνίες αυτές στην ατζέντα σας. Θέλω να σας πω ότι η λήξη προθεσμίας ε, για την γνωμοδότηση ελέγχου προ... προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στις 12. Το χρονοδιάγραμμα μας επιβάλλει ιδιαίτερα ε, στενά χρονικά περιθώρια οπότε σας παρακαλώ οι τροπολογίες σας μόνο στα αγγλικά. Τώρα, η δοτήσεις ε, για τις πανευρωπαϊκές ε, συμφωνίες είναι 22 Σεπτεμβρίου στις 12 και οι σχετικές προθεσμίες θα σας ανακοινωθούν σήμερα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο relativo alla visita della delegazione AFET. Τώρα, Βαν Πρέντα, 8 και 9 Σεπτεμβρίου για την επίσκεψη στην Ισλανδία. Κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε, Μια αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ ε, επισκέφθηκε την Ισλανδία το Σεπτέμβριο. Στην αντιπροσωπεία είχαμε, ήμουν εγώ, η κυρία Κέννη από το ΣΕΛ και η κυρία Τζεντίνη από τους Πρασίνους και η και ο κύριος ο Σερ Ρόμπερτ Άτκινς από, τους, ε, από την ECR. Είχαμε λοιπόν πολύ άσχημο πρόγραμμα για, είχαμε επαφές με δύο υπουργούς, τον ε, Υπουργό Αλληλείας, τον κύριο Γκέμερσον και με τον Υπουργό Ενέργεια, την Υπουργό Ενέργειας και Τουρισμού Επίσης ε, ήρθαμε σε επαφή με τον ε, επικεφαλής ε, για τις διαπραγματεύσεις, τον πρόεδρο του Ισλανδικού Κοινοβουλίου, και με τους εκπροσώπους της Ισλανδικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων καθώς και με εκπροσώπους ΜΚΟ που είναι υπέρ της προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ένωση καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων που είναι κατά της ένταξής της. Εννοείται βέβαια ότι είχαμε επαφή με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, κύριο Σούμα, καθώς και τους πρέσβεις των χωρών μελών της Ένωσης που είναι διαπιστευμένοι στο Ρέγκεβεκ. Τέλος, να φερθώ στην επίσκεψή μας στην ε, γεωθερμικό σταθμό Έλλης, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με διάφορους ειδικού ε, ακαδημαϊκούς από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας για να συζητήσουμε θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, αλλά και η σχέση μεταξύ καθώς και το θέμα της, ε, των περιοχών της Αρκτικής. Να σας δώσω τώρα ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτής της επίσκεψης. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι για μια ακόμα φορά κατανοήσαμε πως έχουμε να κάνουμε με μια υποψήφια χώρα η οποία είναι βαθιά, πολύ βαθιά διχασμένη όσον αφορά την ε, ένταξή της. Δηλαδή, μια χώρα που που πάει σιγά σιγά βλέποντας και κάνοντας είναι το σκεπτικό τους. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του screening και τέσσερα κεφάλαια διαπραγματεύσεων έχουν ανοίξει κατά τη διάρκεια της, ε, της Ουγγρικής ε, Προεδρίας. Δύο από αυτά βέβαια προσωρινά. Θα γίνουν δύο ακόμα γύρι διαπραγματεύσεων υπό την Πολωνική Προεδρία και η φιλοδοξία των Ισλανδών είναι να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια μέσα στον επόμενο χρόνο. Και επίση να κλείσουν αν γίνεται υπό την Δανέζικη Προεδρία. Δηλαδή πολύ φιλόδοξη στόχη. Και θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά τις διαπραγματευτικές τους ομάδες. Οι πυρογνώμονές τους είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και οι εκπρόσωποι της Ένωσης που εργάζονται στην Ισλανδία και έχουν εμπειρία από διαπραγματεύσει, μας είπαν ότι η Ισλανδία είναι σε πάρα πολύ, πολύ καλή θέση από αυτή την άποψη. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα της Ισλανδικής κοινωνίας και των, του, του βαθιού διχασμού όσον αφορά την προσχώρηση της Ισλανδίας. Τώρα, αν και όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ισλανδοί θα πρέπει να εγκρίνουν την προσχώρηση μέσω ρεφερέντουμ, δημοψηφίσματος. Νομίζω λοιπόν πως αυτά τα θέματα είναι ε, πολύ σημαντικά. Υπάρχει γενική συζήτηση ε, σχετικά με ευαίσθητα θέματα. Είναι η αλληλεία, η γεωργία, νομισματικά και το θέμα της Αρκτικής. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά θέματα που προέκυπταν σε όλες τις συναντήσεις και όλες τις συζητήσεις που είχαμε με τις, ε, τους εκπροσώπους της Ισλανδικής κοινωνίας και με τον επικεφαλή της διαπραγματευτικής ομάδας και με όλους ε, τους συνομιλητές. Τώρα όσον αφορά την αλληλεία. Φαίνεται αυτός να είναι, αυτό να είναι το βασικό ζήτημα για λόγω του οποίου η Ισλανδία έχει αναβάλει για τόσο πολύ καιρό την υποβολή αίτησης για προσχώρηση στην Ένωση. Ε, υπάρχει, μέγας, όπως σας είπα, μεγάλη διχόνοια και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. Σα είπα ότι η κοινωνία είναι διχασμένη, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση. Από τη μια πλευρά έχουμε το αριστερό κόμμα, το Ισλανδικό κόμμα, όπως λέγεται, ε, που είναι υπέρ της ένταξη. Το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, το πράσινο κόμμα, που αποκαλείται αριστερό πράσινο κόμμα, ε, είναι ανοιχτά κατά της ένταξη. Και εκείνοι έχουν το Υπουργείο ε, Γεωργίας και Αλίας. Ακόμα ένα κλειδί, ε, χαρτοφυλάκιο κλειδί έχουν οι ίδιοι οι πράσινοι, δηλαδή οικονομίας. Το Υπουργείο Οικονομίας είναι των πρασίνων. Τώρα όσον αφορά τη γεωργία ο Υπουργό Αλληλεία και Γεωργία, ο κύριο Μπιέναρσον, Γιον Μπιέναρσον, που είναι μια από τι κεντρικέ ε, προσωπικότητε του κινήματο κατά τη ένταξη τη Ισλανδία, μα είπε ρητά και ανοιχτά ότι δεν θα δώσει εντολή διαπραγματευτική για τα κεφάλαια της Γεωργίας και της Αλίας ως τμήμα των διαπραγματεύσεων. Και έτσι θα προσπαθήσει να μπλοκάρει τελείως την διαδικασία. Αυτός και άλλοι Ισλανδοί πολιτικοί με τους ίδιους πολιτικούς προσανατολισμούς δημοσία δήλωσαν ότι καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα πριν να αλλάξει η Ισλανδική νομοθεσία στο να υιοθετήσει το κοινοτικό κεκτημένο. Στην ουσία αυτό σημαίνει πως οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διακοπούν άμεσα. Ωστόσο, η Ισλανδική κοινή γνώμη πιστεύει το αντίθετο. Με την έννοια ότι ο κόσμος γενικά πιστεύει πως θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει δηλαδή σύγκρουση απόψεων με τις απόψεις ε, ενός από τα κόμματα που συναποτελούν τον κυβερνητικό συνασπισμό. που όπως σας είπα πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διακοπούν και ότι και η αίτηση που για προσχώρηση της χώρας θα πρέπει να αποσυρθεί. Τώρα, για τα νομισματικά, τα οικονομικά ζητήματα. Πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ισλανδία έχει υποβάλει αίτηση για να μπει στην Ένωση πριν από δύο χρόνια ήταν η κατάσταση της ε, κορώνας, της Ισλανδικής κορώνας που είναι το εθνικό νόμισμα. Όλοι όσοι το συζήτησα μαζί τους ομόφωνα μου είπαν ότι η κορώνα Ισλανδίας είναι πολύ αδύναμο νόμισμα για να μπορέσει να σταθεί στο διεθνές προσκήνιο. Και ότι αν εισχωρούσαν στην Ευρωζώνη θα ήταν αυτό μια μεγάλη ευκαιρία για σταθεροποίηση της Ισλανδικής οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι η Ισλανδική οικονομία μετά από την φρικτή κρίση την οποία διάνυσε πριν από κάποια χρόνια βρίσκεται τώρα σε καλή κατάσταση. Ε, το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη εκεί, έχει μειωθεί δε και η ανεργία. Και το οικονομικό κλίμα εν γέννη είναι καλό. Η μόνη ανησυχία των Ισλανδών πολιτικών έχει αφορά μάλλον τη σταθερότητα του εθνικού νομίσματος της κορώνας δηλαδή και ταυτόχρονα Τέλος να σας πω και δύο λόγια για τη συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους για τις διαπραγματεύσεις ε, υπέρ της ένταξης και κατά της ένταξης. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση διότι μας έδωσε την ευκαιρία να εντοπίσουμε δύο σημαντικά θέματα ότι δηλαδή η συζήτηση περί ένταξης της χώρας στην Ένωση είναι περισσότερο συναισθηματικού τύπου συζήτηση με την έννοια ότι Πολύ λίγα στοιχεία είναι στη υποδιαπραγμάτευση που είναι επίση αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Καταρχήν λοιπόν πρόκειται για συναισθηματικό ζήτημα και όλοι το δέχονται αυτό. Έπειτα είναι προφανές ότι το κίνημα κατά της προσχώρησης είναι πολύ πιο καλά οργανωμένο και δομημένο από ότι το κίνημα υπέρ της ένταξης και υπάρχει σημαντική και ορατή διαφορά όσον αφορά την ε, δέσμευσή τους και την εμπλοκή τους στην διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν την εικόνα που αποκομίσαμε μετά από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ισλανδία και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είμαι πεπισμένος ότι οι διαπραγματεύσει με την Ισλανδία θα είναι ενδιαφέρουσε για τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Ο Σερ Ρόμπερτ Έτκινς, μέλος αντιπροσωπείας της Ισλανδίας, ε, συμμετείχε στην επίσκεψη. Καταρχήν να συγχαρώ τον ε, κύριο Πρέντα για την ε, ηγεσία του στην διαπραγμάτευση. Μας έδωσε στυλ και κύρος ε, και κατά τη διάρκεια που πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και φυσικά ε, μας έκανε να συζητήσουμε και πολύ ωραία και σοβαρά τα θέματα. Συμφωνώ για την κρίση του, για τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Αλίας, ο οποίος μου φάνηκε πως ήταν ε, μόνος και αποκομμένος και από την ίδια την κυβέρνηση και τίποτα στον κόσμο δεν πρόκειται να τον πείσει ότι η ένταξη της χώρας του είναι θετική. Και παρατήρησε μάλιστα όπως και άλλοι πως η Αλία είναι τόσο κρίσιμη για την Ισλανδία, πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε, είναι τόσο σημαντική για την Ισλανδία όσο είναι η λίρα για την ε, Αγγλία. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό μπορεί και να παρεξηγηθεί. Με πάση περιπτώσει, εγώ έθεσα την ερώτηση σε αρκετούς και δεν ε, πήρα ε, οριστικές απαντήσεις. Ε, ε, και είπα, εφόσον υπήρχε τόσο μεγάλη διχόνοια ανάμεσα στα κόμματα, γιατί ε, συνεχίζουν με την αίτηση ένταξης. Και τελικά, σε μια συζήτηση με τον αρχηγό του, αρχη, του κόμματος Ανεξαρτησίας, που είναι το πιο μακρόβιο κόμμα, αν και δεν είναι στην κυβέρνηση, και επίσης του προοδευτικού κόμματος, που είναι το κόμμα ALDE της Ισλανδίας, τους ρώτησα λοιπόν και τους δύο και μου είπαν εγώ είπα δηλαδή που, ότι σκέφτομαι πως ε, η θέση των διαπραγματεύσεων ήταν κάπως αστήρικτη γιατί προχωρούσαν σε μια αίτηση ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε υποστήριξη για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αίτησης. Και ε, τους πρότεινα να ήταν, ότι ήταν πιο λογικό να κάνουν ένα δημοψήφισμα πριν κάνουν την αίτηση που, που πέρασε από το Κοινοβούλιο μόνο με, χάρη σε μία ψήφο, με διαφορά μίας ψήφου. Και χάρη στο γεγονό ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτε και οι πράσινοι, ακόμα και αν οι πράσινοι ήταν αντίθετοι, ήταν έτοιμοι να επιστηρίξουν την ε, αίτηση με μία ψήφο για να μείνει η κυβέρνηση στην εξουσία. Άρα λοιπόν είναι τεταμένη κατάσταση. Εγώ νομίζω λοιπόν πω σπαταλάμε χρόνο και χρήμα με αυτέ τι διαπραγματεύσει, ενώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κ. Πρέντα, ότι δηλαδή η ποιότητα των διαπραγματεύσεων ήταν πολύ καλή, πολύ ψηλή, ότι ο επικεφαλής για τις διαπραγματεύσεις νομίζω πως είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Αλλά λοιπόν όλα αυτά κοστίζουν χρόνο και χρήμα και γιατί τα κάνουμε εφόσον δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Μήπως θα ήταν καλύτερο πρώτα να στηρίξει το Ισλανδικό κοινό την ένταξη και πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και ίσως να γινόταν και ένα δημοψήφισμα για τους όρους των διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής ε, των διαπραγματεύσεων και ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου ήταν αισιόδοξοι και θεωρούν ότι θα, γίνει, θα επιτευχθεί η συμφωνία ακόμα και με το θέμα της αλληλείας ε, έτσι ώστε να έχει ε, τις πιθανότητες να το στηρίξει ο Ισλανδικός λαός. Πάντως ακόμα εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν μπορούμε να το κρίνουμε γιατί εξαρτάται και από άλλα ζητήματα. Δύο παρατηρήσεις όσον αφορά τη δημοσιονομικά, όπως τα συζητήσαμε, όχι με τον Υπουργό, αλλά με τον βοηθό του τα συζητήσαμε. Καταρχήν με εντυπωσίαση που έμαθα ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να μπουν στο ευρώ από ότι να μπουν στην Ένωση εν γέννη. Και όπως ξέρετε οι κανόνες δεν το επιτρέπουν και κάποιοι από εμά που απ' έξω βλέπουμε τα προβλήματα της Ευρωζώνης, Πρόεδρε, που εσείς τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τα μέσα, ε, θα θεωρούμε πως δεν θα πείραζε κιόλα. Ε, επίσης υπέρ τη βρετανική και Ολλανδικής κυβέρνησης οποιαδήποτε κρεμή χρέη που οφείλονται στις οικονομικές τους δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα πριν από ένα-δύο χρόνια θα ξεπληρωθούν πλήρω. και αυτό ήταν ευχάριστη έκπληξη. Κάτι ακόμα, μα ε, γύρισαν, μα γύρισε ένα οδηγό λεωφορείο που στην ουσία ήταν εκπρόσωπο του λαού, ένα Vox Populi, δεν ήταν ένα μέσο ε, οδηγό, ένα οποιοδήποτε τυχαίο οδηγό. Από ό,τι φαίνεται ήταν καθηγητή και έκανε ε, ξεναγήσεις και οδηγού, έκανε τον οδηγό στον ελεύθερο του χρόνου και του είπα μετά από κάθε συνάντηση, μου είπαν ε, αυτά του έλεγα, εσύ τι πιστεύεις και μου έλεγε μπα αυτή είναι όλη πολιτική, μη δίνει σημασία, δεν αντιπροσωπεύουν τον Ισλανδικό λαό και ούτω καθεξής. Τώρα δεν έχω ιδέα αν όλα αυτά λυθεύουν ή όχι, πάντως η αντιπροσωπή μας διασκέδαζε μετά όσα έλεγε ο οδηγός. Υποψιάζομαι όμως ότι ίσως κάποιος πυρήνας αλήθειας υπάρχει σε όσα μας έλεγε. Δηλαδή, ότι πραγματικά κάποιοι είναι υπέρ, αρκετοί κατά και δεν είμαι τελικά βέβαιος αν είναι θετικό ή αρνητικό. Πάντως με εντυπωσίασε η εφημερία που είδαμε και εντάξει μια φωτογραφική εικόνα πήραμε αλλά φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλά. Ο Υπουργό Οικονομικών μας είπε ότι η ανάπτυξη είναι της τάξης του 2% ότι προοδεύουν αλλά στην ουσία Πρόεδρε, προφανώς εξαρτάται από τις διαπραγματεύσει. Αυτή ως δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός δεν έχουν δυσκολία καμία για να συμφωνήσουν με τα διάφορα κεφάλαια, εκτός από τα τέσσερα θέματα που σας ανέφερε ο κύριος Πρέντα και συμφωνώ με την κρίση του. Αν ήθελαμε να μαντέψουμε και η συνάντηση που είχαμε πριν από τη συνεδρίαση με τους πρέσβες όπου πήραμε μια καλή εικόνα για το πώς βλέπουν τα πράγματα είπαν στην ουσία ότι όλα παίζονται στο πλαίσιο της Ισλανδίας δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της αλληλείας υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι κάποιος φρέσκος που έρχεται στην κοινή αλληλευτική πολιτική δεν θα ήταν και τόσο άσχημο και κατά συνέπεια θεωρώ ότι τελικά μπορεί διστακτικά να ψηφίσουν υπέρ της ένταξης Έστω και αν γίνει μόνο και μόνο για τα θέματα νομισματικά, γιατί το νόμισμά τους είναι ένα μικρό και αδύναμο νόμισμα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη Γραμματεία ξανά και τον αρχηγό της αντιπροσωπείας που με πολύ στυλ και χιούμορ ε, ολοκλήρωσε την αποστολή. Ε, ευχαριστώ κύριε Άτκινς. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της αντιπροσωπείας για την ενημέρωση αυτή και την επισκέψη την ίδια. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω ότι είχα την ευκαιρία εν τω μεταξύ να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο και φαίνεται ότι θεωρεί πως η, Ιρλανδ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρόπον την να προδώσει την Ισλανδία. Όταν κάποιες ασιατικές χώρες ε, είδαν περισσότερη προσοχή να δίνεται και στήριξη σε περίπτωση κρίσεως, ε, Φερρυπίν, ε, αναφερόμενος ή λίγο πολύ έχοντας το μυαλό του σε στήριξη προερχόμενη από την ε, Κίνα και σχέσεις Κίνας-Ισλανδίας. Βλέπει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοήθησε τόσο. Επίσης φαίνεται ότι στο Ρέικεβικ θα δοθεί εντολή στην αντιπροσωπεία να ε, μπλοκαριστούν τα θέματα της, ε, των διαπραγματεύσεων στην Αλία Ίσως λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε την πρότασή τους για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την ε, ε, προβολή της Ισλανδίας σαν ε, ακρογωνιαίου λίθου για την αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα αρκούν για να τους πείσουν. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε Τάραντ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο Βόκτορ Γκρίπα από την Υπηρεσία Εξωτερικών. Ευχαριστώ. Ακούσαμε με ενδιαφέρον την έκθεση του εισηγητή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και αντιστοιχούν με τις πληροφορίες που έχουμε στην υπηρεσία εξωτερικών. Εμείς θα μελετήσουμε τις εξελίξεις της Ισλαμικής εσωτερικής πολιτικής και θα προσέξουμε ιδιαίτερα την πολιτική της Αρκτικής. Πρόκειται για μια κοινή πολιτική που εμπλέκει την Ισλανδία, την Νορβηγία και τη Ρωσία. Οι εξωτερικές μας υπηρεσίες ασχολούνται με το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ δόκτωρα Γκρίπα. Παρακαλώ κύριε Άτκινς. Ε, πρόεδρε, με συγχωρείς, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ακόμη και το λησμόνισα πριν. Αλλά ύστερα από αυτά που ακούσαμε, ο κύριος Νταμπρέιντα είπε κάτι για την ε, Αρκτική και θέλω να το υπογραμμίσω ότι φαίνεται πως υποψιάζονται πως την Ισλανδία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούν θεωρούμε την Αρκτική πιο σημαντική από την Ισλανδία και από την άλλη και εκείνοι πιστεύουν ότι με την ένταξή τους μπορούν να, είναι πιο, να καταστούν πιο ισχυροί στην, στην, στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα, εν προκειμένου η Αρκτική, το οποίο πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία να χειριστούμε, διαφορετικά θα φέρει αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λαμβάνουμε υπόψη μας ε, το μήνυμά σας προς την Κομισιόν και θα το, θα το γράψουμε και στα πρακτικά. Πάμε τώρα στο σημείο 4, αλλά είπαμε στο 4 θα εξετάσουμε την έκθεση Λίζεκ για για τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Τώρα, την ε, αναθεώρηση της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής γειτονίας θα τη συζητήσουμε στο 5 για να μπορέσει να συμμετέχει ο κύριος Μπρόκ. Θα τη συζητήσουμε είπαμε 10 και 4. Το σημείο της κυρίας Νίλσεν θα πάει τελευταίο. Ο κύριος Λίζεκ. Παρακαλώ. Η κυρία Λίζεκ. Δεν κυρία. Δεν κυρία. Ναι. ναι, πρόεδρε, αλλά πρέπει να πω ότι βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια ε, και δεν βλέπω, με την κυρία δεν έχω συνοηθεί τίποτα, δεν καταλαβαίνω τι μου ζητάτε. Ούτε κι εγώ σήμερα το πρωί το έμαθα. ότι ο κύριος Μπρόκ είχε διάφορες δεσμεύσεις και προσπάθησα να συνδυάσω τα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ίσως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα άλλο κριτήριο. Εντάξει, πρόκειται για κυρία βέβαια. Αλλά οι σκεώδεις εισηγητές έχουν... μία βαθμίδα λιγότερο από έναντι των επισήμων εισηγητών. Λοιπόν, κύριε Λιζεκάν, είστε σύντομος, θα έχουμε χρόνο για όλα φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι. Λυπούμε που εξαιτία μου αλλάξαμε τα σχέδια της κυρίας Γέγκλερ. Ζητώ συγγνώμη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, γιατί εξάλλου έχετε μπροστά σας το σχέδιο έκθεσης και επιτρέψτε μου απλώς ε, να σας ε, υποβάλω μία προσωπική παρατήρηση. Όταν με διορίσατε εισηγητή ήμουν πανευτυχής, αλλά συνειδητοποίησα αμέσω ότι το έργο μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή το θέμα της γεωργίας δεν είναι καθόλου απλό και ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να, να συντάξω την έκθεσή μου για τη γεωργία και να λάβω υπόψη μου όλες τις ε, πτυχές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές ε, συνιστώσεις που αποτελούν αυτή τη χώρα η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι πολίτες αυτής της χώρας ονειρεύονται κάποια μέρα να γίνουν μέλη της Ένωσής μας. Πήγα τρεις φορές στη Γεωργία όταν ετοίμαζα την έκθεση και τρεις φορές συνάντησα τόσο τον πρόεδρο της χώρας, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της ε, Γεωργίας και με τους ε, πολιτικούς ε, της αντιπολίτευσης που βρίσκονται εκτός Κοινοβουλίου. Μίλησα με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με τον διαμεσολαβητή, με τους δημοσιογράφους, με όλους όσους ασχολούνται στην ε, Γεωργία με, τα με διάφορα θέματα που αφορούν σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μίλησα με Γερμανούς, με Άγγλους, Πολωνούς κτλ. Μίλησα με τον κύριο Μπριγκάντα που είναι ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Γεωργία και τους συνεργάτες του. Έλαβα πολύ χρήσιμες πληροφορίες πληροφορίες για το ποια είναι η οικονομική κατάσταση στη Γεωργία μετά από τη σύραξη με τη Ρωσία το 2008. Αυτά τα οποία έγραψα στην έκθεσή μου καταδεικνύουν ότι η Γεωργία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, και για τον εκδημοκρατισμό οι εκλογές, οι περασμένες εκλογές εκτελήχθηκαν πάρα πολύ ομαλά αυτό το διαπίστωσαν ε, και οι παρατηρητές που συμμετείχαν στην διαδικασία έχουμε πάρα πολύ γρήγορη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Γεωργία και στη θεσμική μεταρρύθμιση. Υπάρχει βέβαια ένα πολιτικό, ένα πολιτικό πρόβλημα που είναι και το αποτέλεσμα του πολέμου το 2008. Πρόκειται για μία κατάσταση που πρέπει να καθοριστεί σαφώς. Το 20% της επικράτειας της Γεωργίας σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι κατεχόμενα εδάφη. Εμείς, η διεθνής κοινότητα, πρέπει να αναγνωρίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της γεωργίας και διαπιστώνουμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα στην επικράτεια. Ένα άλλο θέμα είναι η συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. Θεωρούμε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για το σεβασμό των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και να βοηθήσουμε τους γεωργιανούς μας εταίρους να μεταρρυθμιστούν. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ήδη συζητήσα, ε, ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές ε, και είμαι έτοιμος να ακούσω όλες τις παρατηρήσεις. Η ε, κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση που σεβάστηκε και το όλο χρονοδιάγραμμα. Είχαμε χρόνο και για διαβούλευση, για συζήτηση. Τον ευχαριστώ. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν ε, ε, μεγάλες δυσκολίες ε, στην έγκριση αυτού του κειμένου. Πρόκειται για ένα κείμενο πάρα πολύ ισορροπημένο. Καλύπτει τα κύρια προβλήματα της προόδους αλλά και τα κενά. Έχουμε κοινέ αξίες με την γεωργία, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και οικονομική ανάπτυξη, όπως είπε και ο κύριος Λίσεκ, τα, είναι τεράστιες οι πρόοδοι της Γεωργίας. Όμως ε, το κράτος ε, θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Πλουραλισμός ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην πολιτική. Πρέπει να προχωρήσει στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης χρειάζεται, τονίζουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα εθνικής κυριαρχίας του Γεωργιανού κράτους και πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσφύγων από την Νότια Οσετία και από την Απκαζία, Απκασία έχουμε κινήσεις πληθυσμών που αμφισβητούν κάθε φορά τα σύνορα, τη γραμμή των σύνορων. Καλούμε κατά συνέπεια τη, Γεωργινή, τη γεωργιανή κυβέρνηση να μην προσφεύγει στη βία για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το θέμα της χορήγησης θεωρήσεων επίσης πρέπει να εξεταστεί και να οδηγηθεί προς μία απολευθέρωση. Όμως έχουμε και μερικές αμφισβητήσιμες πολιτικές κινήσεις. Παρά την κάπως περίεργη ανεξαρτησία των ομόρων χωρών της Γεωργίας, η Γεωργία πρέπει να προχωρήσει στο δρόμο της. Να αποφεύγει την αστυνομική βία. Πρέπει να προωθήσουμε τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να δούμε το θέμα των φυλακών και τις συνθήκες κράτησης μέσα σε αυτές τις φυλακές οι οποίες ε, υποφέρουν από υπερπληθυσμό. Η Ένωση Συντακτών της Γεωργίας επίφθινε μία έκκληση για την Νότια αιτία όπου κρατείται ένα Σέρβος δημοσιογράφος ε, με την κατηγορία ότι είναι κατάσκοπος της Ρωσίας. Εχθές είδαμε και ένα φωτορεπορτάζ σχετικά με δημοσιογράφους οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Χρειάζεται ελευθεροτυπία. Χρειάζονται, χρειάζεται οι δημοσιογράφοι να έχουν πρόσβαση στις πηγές. Κάτι πρέπει να κάνει η Γεωργία προς αυτήν την κατεύθυνση όπως έλεγε και ο κύριος Λίσεκ. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι η Γεωργία βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Ο κύριος Μπροκ. Πρόεδρε, μερικές παρατηρήσεις θα ήθελα να διατυπώσω. Και συνεχίζω εκεί που σταμάτησε η προλαλή Ότι δηλαδή η Γεωργία έχει μπει στο σωστό δρόμο και ότι δεν έχουν βεβαίως όντως επιτευχθεί όλα όσα θα θέλαμε 100% αναμενόμενο άλλωστε. Πλην όμω, μετά τον πόλεμο, βλέπουμε ότι η γεωργία έχει μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να βελτιώσει την οικονομική τη κατάσταση, να αναπτύξει τι υποδομέ τη, να εξυγχρονιστεί, να έχει καλού δείκτε ανάπτυξη και έχει καταφέρει να εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα πριν από μερικά χρόνια να περιμένω εγώ. Όταν λοιπόν τον Νοέμβριο πήγαμε συναδέλφους ε, στην ε, Γεωργία ως παρατηρητής μαζί με άλλους ε, και από το Κοινοβούλιο και από τους εθνείς παρατηρητές για τις δημοτικές εκλογές, για τις τοπικές εκλογές, διαπίστωσα ότι αυτές εξήχθησαν κανονικά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει τη χώρα να την υποστηρίξουμε στην προσπάθειά της να συνεχίσει τον δρόμο που έχει πάρει. Άλλωστε επισημαίνω ότι υπάρχουν άλλες χώρες από την Ανατολική γειτονία που δεν έχουν να επιδείξουν τόσο καλές επιδόσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Χωρίς όμως και να παραμελήσουμε την υπόδειξη κάποιων πιο αδύναμων σημείων και την ανάγκη να, ε, ανάγκης μάλλον να ε, εξασφαλιστούν πρόοδοι και βελτιώσεις στα αδύναμα αυτά σημεία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Δόκτωρ Γιάερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ που προσκαλέσατε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να σας παρουσιάσει τις απόψεις της στην υπόθεση αυτή. Εάν μου επιτρέπετε θα ήθελα ένα δύο λεπτά να μείνω, να σταθώ στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Έχουμε μέχρι στιγμή διεξεγάγει 7 συνόδου ολομελία. Τελευταία διορθώνει ο ομιλητή 6, τελευταία ήταν τον Ιούλιο και η 7η προβλέπεται για τον Οκτώβριο. Τώρα έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στους περισσότερους των τομέων. Κάποια ζητήματα παραμένουν εκκρεμή, είτε επειδή έχουν κάποιο διάζοντα σχέση με τη γεωργία χαρακτήρα, είτε γιατί είναι ζητήματα τα οποία γνωρίζουν ως ε, δυσκολίες και άλλοι εταίροι κατά, τον, κατά αντίστοιχο τρόπο. Πάντως πρόοδο σημειώνεται και θα ήθελα να σημειώσω ότι είχαμε επαφές και ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές πριν από τις θερινές διακοπές. Ελπίζω ότι μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία αυτής της εκθέσεως. Ε, υπευλήθη σχέδιο εκθέσεως το Σεπτέμβριο σε, στην υπηρεσία μας για σχόλια και αν μου επιτρέπετε τώρα για την έκθεση αυτή θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να συνεχίσω ε, με σχόλια για κάποιες από τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων σας. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πως η Γεωργία έχει προχωρήσει σε αξιόλογες μεταρρυθμίσεις και σε βάθος αλλά και ταχαίως. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχουν φτάσει στο στόχο τους ακόμα οι γεωργένοι. Εμείς έχουμε επισημάνει στην έκθεση πρόοδου ε, δύο ζητήματα στα οποία θα θέλαμε να δούμε πρόοδο. Το ένα είναι η εδραίωση της δημοκρατίας και η εξασφάλιση πολιτικού κλίματος, πολιτικής νοοτροπίας, ανοχής της διαφοράς και πλουραλιστικής θα την ονόμαζα και το άλλο έχει να κάνει με την ελευθερία των μέσων μαζική που υπεγράμψει και κάποιος από τους συναδέλφους νωρίτερα και που έχουμε και εμείς ιδιαίτερα τονίσει. Προσπαθούμε τα θέματα αυτά βεβαίω να τα επαναφέρουμε και να τα προβάλλουμε στι διαπραγματεύσει και μέσα από τη συνεργασία μα με τι αρχέ τη Γεωργία. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το θέμα του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας. Διατυπώνετε εσείς εδώ κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς ε, προκύπτει η παραπομπή στο άρθρο 49 της συνθήκης, σαφώς ε, ως σημείο εμφανές της εκθέσεώς σας. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω τη συμφωνία σύνδεσης που διαπραγματευόμαστε εμείς με τους εταίρους μας οι συμφωνίες σύνδεσης δεν προϋποθέτουν αυτές καθεαυτές ούτε και αποκλείουν η αδίποτε μελλοντική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποτελούν μόνο συμφωνίες πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης χωρίς να αποκλείουν καμιά περαιτέρω εξέλιξη. Και επίσης θα να υπογραμμίσω ότι όταν γίνεται η διαπραγμάτευση τέτοιου είδους συμφωνίες πως ε, εκ παραλίλου προχωρούν και ε, σχετικές φιλοδοξίες ή βλέψεις των εταίρων μας προς την κατεύθυνση αυτή. Για τις ε, περιοχές τώρα, αυτονομημένες περιοχές Απχασίας και ε, Νότιας Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, όπω έχει υπογραμμίσει πολλέ φορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνεται σεβαστή η εδαφική αικαιρότητα τη Γεωργία. Αυτό το υπογραμμίζουμε τακτικά. Και αυτή είναι και η βάση τη προσεγγίσεω την οποία ακολουθούμε προκειμένου να χειριστούμε το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να επισημάνω ότι αξιοποιούμε μια σειρά μέσων, ευρύ φάσμα μέσων, όπως τη ε, διαδικασία της ε, Γενέβης, ε, τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, τον ειδικό ε, πεσταλμένο που πρόσφατα διορίστηκε, την ε, στήριξη στους εσωτερικά εκτοπιστέντες, την υποστήριξη για την οικονομική ε, ανάπτυξη, μέσα τα οποία ήδη αναφέρονται και στην έκθεσή σας. Και θα ήθελα για τις συστάσεις σας, αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ο μηχανισμός παρακολούθησης η UMM θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί όπως έχει τώρα ε, για να παρακολουθεί την κατάσταση και από τις δύο πλευρές του διοικητικού συνόρου. Και για τις αυτονομημένες περιοχές πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση πάντα με σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας ε, έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε σε να μην προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναγνώριση των περιοχών αυτών, των εδαφών αυτών, αλλά και να μην τις απομονώσει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε ε, συνθήκες πιστεύω με τον τρόπο αυτό για μια μακροπρόθεσμη αλλά και ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Για τις ε, διαπραγματεύσεις στη, της Γενέβης για τις οποίες διαγιγνώσκω μια απεσιόδοξη τάση και κρίση στην εκθεσή σας πιστεύω θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αποτελούν το μόνο φόρουμ αυτή τη στιγμή επαφής μεταξύ των πλευρών και επιπλέον των αποτελεσμάτων που και εσείς επισημαίνετε η ίδια η διαδικασία της Γενέβης παραμένει σημαντική αυτή καθεαυτή και γι' αυτό και την υποστηρίζουμε θερμά. Επίσης, για τη διαδικασία διευκόλυνσης και επανεισδοχής, διευκόλυνσης θεωρήσεων διαβατήριου και επανεισδοχής που έχει τηθεί πλέον σε ισχύ. Θα έλεγα ότι πριν αναλυφθούν περαιτέρω βήματα για να εμπαθυνθεί αυτή η συνεργασία, ενίσχυση της κινητικότητας δηλαδή, θα πρέπει να καταγράψουμε κάποιες καλές επιδόσεις τόπου, Θα έλεγα δηλαδή ένα χρόνο μετά τη θέση ισχύ αυτής της συμφωνίας να την επανεξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις συνθήκες υλοποίησης της. Για δε την ε, ίδια την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, ε, θα είναι ασφαλώς συστατικό τμήμα μια συμφωνία σύνδεσης και σημαντικό. Πιστεύω ότι φτάνουμε πλέον στο τελικό στάδιο των προπαρασκευαστικών μας ε, προσπαθειών. Έχουμε συμφωνήσει με τις αρχές της Γεωργίας σε ένα πολύ σαφές σχέδιο δράσεως, το οποίο τώρα, ε, στο οποίο τώρα ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εφαρμογής οι αρχές, Πρόγραμμα δράσης που ολοκληρώνεται λοιπόν στο σχεδιασμό του και του οποίου την θετική αξιολόγηση έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες της Επιτροπής έτσι ώστε να είμαστε θέσει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που έχω θα ήθελα τις παρατηρήσεις μου να τις περιορίσω σε αυτά τα Ευχαριστώ πολύ, αλλά πολύ ευχαριστώ να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Γιάιρ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και λυπούμε που δεν ήρθα νωρίτερα. Είχα ένα πρόβλημα ερχόμενοι εδώ. Σας ευχαριστώ πάντως και θα ήθελα Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσεκ για την πρόταση που έκανε και το σχέδιο που έχει συντάξει. Να αναφέρω κάποια θέματα όπου θα υποβάλουμε τροπολογίες γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπως πιο ανοιχτή, δηλαδή να δούμε τις διάφορες πλευρές των προβλημάτων. Συμφωνία σύνδεσης με τη Γεωργία. Από τη δική μας πλευρά, από ό,τι θυμάμαι, τέσσερις φορές γίνανε συγκρούσεις και αναφέρεται η ρωσική κατοχή κτλ. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό και εγώ το επικρίνω, αλλά θα πρέπει να το διατυπώσουμε με κάποιο τρόπο που να αφήνει το δρόμο ανοιχτό ώστε να μπορέσουμε μαζί με τους, τον ΟΗΕ επιτόπου και να, να δουλέψουμε στα κατεχόμενα εδάφη, να βρούμε τρόπο δηλαδή να βοηθήσουμε τον κόσμο τέτοιο είδους τροπολογίες θα καταθέσω. Ε, επίσης υπάρχει μια τροπολογία όπου κάνετε λόγο για την επικοδομητική μονομερή προσέγγιση που την ε, καλωσορίζεται και το ενομιλία του Προέδρου Σακασβίλη όταν ήταν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι. Ωστόσο, εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την πρόταση του Συμφώνου για μη επίθεση πράγμα που είχε ξεκινήσει πριν από την ρωσική εισβολή το 2008 και τότε η ε, Γεωργία και ο Σεκασβίλη δεν θέλαν να το δεχτούν Νομίζω λοιπόν πως έχει νόημα να το αναφέρουμε. Για το TCFTA εμείς όπως μπορείτε να φανταστείτε θα θέλαμε να γίνει ένας, μια αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου πριν να ξεκινήσει. Γιατί όπως έχουμε δει με άλλους υπάρχουν πάντοτε προβλήματα, ιδιαίτερα για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να αναφέρω και ελπίζω πως θα βρούμε κάποια συμφωνία. Σας ευχαριστούμε κυρία Λούνα Τσέκ. Τελικά σχόλια από τον εισηγητή, τον κύριο Λίζεκ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για όλα τους τα σχόλια σκιώδεις συγητές, ε, τον εκπρόσωπο Τη υπηρεσίας εξωτερικών. Είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε συζήτηση, θα τα βρούμε σίγουρα και θα συμφωνήσουμε. Πολύ ωραία κύριε Λίζεκ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 28 Σεπτεμβρίου στις 12. Όπως είπα και πριν, πάμε τώρα στο σημείο 7. Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ο κύριος Μπροκ έχει το λόγο πρώτος για την νότια πλευρά. Ο κύριος Δαβίδ, ο συνεισηγητής, σήμερα δεν θα είναι παρόν. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μπροκ. Ο κύριος Μπροκ δεν ακούγεται. Μάλιστα. Τώρα με ακούτε. Έχω την τιμή να παρουσιάσω ε, εκ μέρους του κυρίου Νταβίτ ε, μία έκθεση για το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ιδιαίτερα με έμφαση στην νότια γειτονία ελπίζοντας ότι ε, σημειώνοντας μάλλον ότι πρέπει να ε, δοθεί η νέα εστίαση στην ε, πολιτική γειτονία αλλά και ελπίζοντας ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εδώ εκπροσώπους της θα δούμε μία νέα προσέγγιση. Πρέπει εδώ να πάρουμε νέες οδούς, νέους δρόμους και μην ξεχνάμε ότι το αραβικό air μας έχει δώσει και νέες δυνατότητες για ε, νέα προσέγγιση. Η πολιτική γειτονίας όμως ε, πλήττεται και από τα οικονομικά προβλήματα, τα δημοσιονομικά προβλήματα που σοβεί και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε πρόσφορα μέσα ώστε αυτή η πολιτική γειτονία να στηρίξει τα αραβικά αυτά κράτη, τα γειτονικά μας κράτη, στο δρόμο τους για τη δημοκρατία, το δρόμο που επιδιώκουν χάρη σε αυτές, επιδιώκουν να επιτύχουν χάρη σε αυτές τις επαναστάσεις. Το δρόμο σε τελευταία ανάλυση τον οποίων ε, διεκδίκησαν και ε, πήραν τελικά τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πριν από δύο δεκαετίες. Μπορούμε λοιπόν να ε, στηρίξουμε τα κράτη αυτά με καλύτερη εστίαση των κονδυλίων που διαθέτουμε, με την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος ή καταπιστεύματος καλύτερα για την ε, δημοκρατία, European Endowment for Democracy, και με ιδιαίτερη έμφαση σε μέσα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο ε, μου προσφέρει ιδιαίτερη χαρά. Η ιδέα δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο καταπίστευμα. Υπάρχουν κονδύλια, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο δεν αξιοποιείται από ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι ποσά αυτά τα οποία θα μπορούσε να, αξιοπο... να αξιοποιήσουν η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και μάλιστα παρά τη θέληση κάποια κυβέρνηση ε, στον αγώνα ακριβώ για την ελευθερία και τα ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αν μπορούσαμε να αναπτύξουμε αυτό το European Endowment for, um, Endowment for Democracy θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τα κράτη αυτά. Πρώτον αυτό λοιπόν. Δεύτερον, σημαντικό είναι να καταστήσουμε σαφές τα κράτη αυτά ότι στηρίζουμε, βοηθούμε τις προσπάθειές τους για τη δημοκρατία και ότι η ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών ε, όπως σε παραδείγμα τη διεξαγωγή ελεύθερων και ανώθευτων εκλογών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης στην έκθεση ο συνάδελφος αναφέρεται σε ορισμένα ζητήματα όπως μετανάστευση, στήριξη της αγοράς εργασίας, κινητικότητα κτλ. Και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία, συνεργατικές σχέσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, του τομέα δηλαδή της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής, που μπορούν με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουν ε, σε μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στον χώρο της Νότιας Μεσογείου. Και ακριβώς ε, ο οικονομικός αυτός χώρος Ευρώπης ε, Νότιας της Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει και μία εναλλακτική οδό επαφής για τα κράτη αυτά, τα οποία έχουν μείνει σε παλαιές οδούς απεικιοκρατικών σχέσεων, εμπορικών απεικιοκρατικών σχέσεων και τα οποία πιστεύω θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και με κίνητρα να αναζητήσουν νέες ε, οδούς εμπορίου, νέες εμπορικές σχέσεις και μεταξύ τους Πράγμα το οποίο βέβαια θα ειστερίξει όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς να υπάρξει αυτή η περιφερειακή ε, διασύνδεση και συνεργασία δεν νοείται. Στη τελευταία ανάλυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ε, συνεργασία με το σκοπό την εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων ε, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε και στη σχέση μας με τα ε, κράτη της Νότιας Όχθης Μεσογείου στην Νότια Γειτονία. Όπως είπα λοιπόν, εδώ είμαι αναπληρωτής ε, εισηγητής. Πιστεύω ότι η έκθεση εκφράζει τις θέσεις των, ε, και των ε, λοιπόν ε, συναδέλφων. Θα ακούσω τις παρατηρήσεις τους φυσικά Είμαι βέβαιος όμως ότι και ο κύριος Δαβίτ ε, θα ε, ακούσει με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις που θα του διαβιβάσω. Θα τις λάβει υπόψη και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που πρέπει να καταθέσει την έκθεση, αν δεν απατώμε... 7 ε, Οκτωβρίου πρέπει να κατεθεί η έκθεση. Μέχρι τις 7 λοιπόν είναι διατεθειμένος να λάβει υπόψη όποιες τροπολογίες έχουν οι συνάδελφοι στο κείμενό του, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της, της ε, εκθέσεως με όσο δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία. Θα ήθελα να σημειώσω ότι τις, ε, το τελευταίες προάλλες που είχα πάει σε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο αισθάνθηκα οργή και αγανάκτηση ακούγοντας ότι πολύ μεγάλα ποσά και ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό της βοήθειας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, χώρα αυτή και ποσοστά 60-70% των κονδυλίων δαπανώνται για μελέτες και μόνο. Μελέτες λοιπόν και όχι έργα. Εγώ ε, ξέρω το λάθος αυτό το είχαμε κάνει και στο παρελθόν με την Ανατολική Ευρώπη, ελπίζω να το επαναλάβουμε. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η υπόθεση και να δώσουμε τα λεφτά εκεί που πραγματικά χρειάζονται στην πράξη και στην, ε, σε ουσιαστικά και πρακτικά σχέδια και όχι σε μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπρόκ. Για το βόρειο τμήμα Έπρεπε να μας μιλήσει ο κύριος Σίβιτς, αλλά δυστυχώς λείπει. Αν θέλουν ε, οι συνάδελφοι να σχολιάσουν τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μπρόκ, ε, έχουμε χρόνο και ξεκινάμε τη συζήτηση. Ο κύριος Μίλαν μόνο. Ε, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ λυπάμαι γιατί έφτασα λίγο αργά γιατί νόμιζα πως ε, αυτή η συζήτηση θα γινόταν ε, κατά τις 12 ε, υποτίθεται, ε, αλλά την φέρατε πιο νωρίς. Άκουσα την παρέμβαση του κυρίου Μπρόκ και εντάξει εν γέννη είναι πολύ καλή έκθεση και πιστεύω ότι προχωρεί, όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ, προς τη σωστή κατεύθυνση. Λυπούμε μόνο που δεν την διάβασα με τόσο πολύ προσοχή όπως θα έπρεπε. Ωστόσο θα ήθελα να κάνω τρεις αρχικές παρατηρήσεις που μου ε, Ήρθα στο μυαλό με τη βιαστική αυτή ανάγνωση που έκανα του κειμένου. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι για ολόκληρη τη Μεσόγειο θα έπρεπε κάπως να βελτιώσουμε την αναφορά στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Πιστεύω πως είναι ένας ε, φιλόδοξος πολιτικός στόχος, είναι μια φιλόδοξη, ένας φιλόδοξος θεσμός και ότι αυτό σχετίζεται με τις προσπάθειες και τα συγκεκριμένα περιφερειακά προγράμματα δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την ιδέα και να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, το τμήμα που αφορά τις ε, συμφωνίες σύνδεσης, στην παράγραφο 13 λέει ότι αναφέρεται στο εμπόριο. Εγώ ήθελα όμως να, εκτός από το εμπόριο να μιλάμε και για τις υπηρεσίες. Εδώ δεν φαίνεται πουθενά η λέξη υπηρεσίες, εκτός από το εμπόριο δηλαδή. Να μην ευνοείται μόνο μία ερμηνεία ε, αγαθών ή προϊόντων. Θα ήθελα να υπάρχει και η λέξη υπηρεσίες και θα το κάνω μέσω μια. Ε, θα το προτείνω μέσω μιας τροπολογίας. Και έπειτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν, δεν πρέπει να ανοίξει μόνο αυτή την αγορά Θα πρέπει το άνοιγμα να είναι αμφίδρομο. Και η Ένωση να ανοίξει λέει κατά συνέπεια το εναγορά τη, αλλά θα πρέπει να είναι όπως σα είπα αμοιβαίο το άνοιγμα. Στην ε, θέμα αυτό οι υπηρεσίε μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί οι υπηρεσίε πιο εύκολα μπαίνουν στις αγορές. Ε, τελευταία μου παρατήρηση και τελειώνω πρόεδρε γιατί δεν πάμε πολύ καλά από χρόνο. Όλο το θέμα αυτό που αφορά την κινητικότητα. Ε, η Ένωση πρέπει να βελτιώσει το θέμα της μετανάστευσης, ε, η διακή προσοχή να δώσει στους νεότερους ε, κτλ. κτλ. Και όσον αφορά το θέμα των μεταναστευτικών ροών, η συνεργασία των τριών χωρών είναι απαραίτητη. Ε, δεν ε, μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο μερός τις ροές. Οι τρίτες χώρες, οι γειτονικές χώρες θα πρέπει και εκείνες να παίξουν ρόλο. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και σε αυτό το θέμα κάπως να διορθώσουμε τη διατύπωση και το θέμα της εισδοχής των μεταναστών θα πρέπει να έχει πιο ξεχωριστή θέση στο κείμενο. Τίποτα παραπάνω, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μίλαν Μόν. Εν τω μεταξύ έφτασε και ο κύριος Σίβιτς που είναι εισηγητής για το βόρειο τμήμα της γειτονία και στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Ε, ε, θα ξέρετε ε, πως η έκθεση αυτή είναι μόνο ένα από τα πολλά σημεία μέσα στην αναθεώρηση της ε, πολιτικής γετνίασης. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση επί του θέματος και γι' αυτό θα περιορίσω τα σχόλιά μου στα συμπεράσματα της έκθεσης. Ε, γιατί η έκθεση αυτή στόχο έχει να ολοκληρώσει την αναθεώρηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ε, γεγονός μάλλον, στο οποίο θα συμμετέχουμε, είναι η διάσκεψη κορυφής της Ανατολικής ε, Εταιρικής Σχέσης στη Βαρσοβία, όπου και εκεί θα περιμένουμε κάποια συμπεράσματα που θα εμπλουτίσουν το τελικό κείμενο της έκθεσης. Εγώ θα ήθελα να δείξω τρία θέματα που είναι πολύ σημαντικά και που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμή στην έκθεση. Καταρχήν, η έκθεση είναι εξαιρετικά συνεκτική με το θέμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής, διότι δείχνει πάρα πολύ καλά όλα τα νέα στοιχεία πίσω από την ε, νέα πολιτική ε, Σε Θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και είχαν ε, ήδη αναφερθεί σε παλιότερα ε, κείμενα της Κομισιόν. Δεύτερον, τώρα αυτά περιλαμβάνονται στην ίδια τη δομή της έκθεσης και θέλουμε να εξασφαλίσουμε την συνοχή ανάμεσα στην Ανατολή και τον Νότο είναι σαφέ πω δεν πρόκειται για, μια, για δύο ξεχωριστέ εκθέσει, μία για την Ανατολή και μία για τον Νότο. Είναι μία ενιαία έκθεση που αναφέρεται σε μια κοινή ε, πολιτική γυμνίαση. Τρίτο σημείο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε περαιτέρω να διαχωρίσουμε σε υποσημεία, συγκεκριμένες δηλαδή αναφορές. την αρχή του περισσότερα για, τα, για περισσότερα ή έτσι ώστε η τα συγκεκριμένα σημεία απαιτήσει ε, θα πρέπει να ε, υιοθετηθούν από τους εταίρους μας, να δημιουργήσουν δηλαδή το δικό του σενάριο για τις αναπτυξιακές πολιτικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει σύμφωνα με το πώς είναι έτοιμη να συνεργαστεί ενώ εφαρμόζει την πολιτική όπως έχει ε, προγραμματιστεί. μία συνθήκη, μία προϋπόθεση πρέπει να τονιστεί. Επίσης θα πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη στιγμή για την κατάργηση των θεωρήσεων, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό από πολιτικής άποψης και για την οικοδόμηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στους πολίτες αυτών των χωρών. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ επίμαχο και, θα, και ήδη ε, φαντάζομαι επειδή είναι κοντά μου κάθεται ο κύριος Μπρόκ ε, ότι αυτή το, η αντιπεράθεση θα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή να τεθεί το θέμα της ένταξης ή όχι στην έκθεση. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σίβιτς και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Σβάλτς που είναι σκιώδης εισηγητής. Ein όχι Σολτς. Με ε, ε, Y, όχι με περιπτώσει, ε, μια γραμμούλα μπορεί να αλλάξει όλη τη φωνητική, όλη την προφορά του ονόματος. Λοιπόν, βλέπω ότι εδώ έχουμε μια καλή έκθεση, μια ε, ε, πλήρη έκθεση με θετική προσέγγιση στα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και προσέγγιση αντίστοιχη με αυτήν την οποία και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ιδιαίτερη έμφαση πάντοτε υποστηρίζουμε. Αυτό που θα ήθελα λίγο περισσότερο να δω και απαιτώ θα έλεγα μάλιστα να αλλάξει είναι στο θέμα αυτού ε, ιδρύματος, του καταπιστεύματος για τη δημοκρατία να έχουμε πιο συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για το τι ρόλο θα διαδραματίσει, τι είδους πρικοδότηση θα έχει, τι καθήκοντα θα αναλαμβάνει το ίδρυμα αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε ποιο βαθμό θα μπορεί ή θα διαδραματίζει κάποιο ρόλο αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε διαφορές διεθνής ε, στο μέλλον. Όπω σε παράδειγμα στην περίπτωση Λευκορωσία, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, προβλήματα και τριβέ σε σχέση με την εκλογή, με τι προεδρικέ ε, εκλογέ. Επίση στη Τρανσνιστερία. Θα έχει κάποια θέση ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επίλυσης των διαφορών η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι θα θέλαμε να ενισχύσουμε τι δυνατότητε που μπορεί να έχει η κοινωνία των πολιτών. Ήδη από το Φόρουμ Κοινωνία των Πολιτών ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ανατολική Γειτονία Ανατολική Εταιρική Σχέση καλύτερα. Είχαμε πολύ καλή εμπειρία, κυρίως από τη Λευκορωσία, ε, από τη Euronest, ιδέα οι δέκα εκπρόσωποι της Λευκορωσίας δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν, έμειναν κενά τα έδρανα ε, που τους είχαμε ε, κρατήσει. Ελπίζουμε όμως να είναι πιο δημοκρατική η κατάσταση του χρόνου και να τους δούμε. Πέραν λοιπόν της Λευκορωσίας έχει προχωρήσει καλά αυτή η συνεργασία. Και θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους εξελίξεις και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι θεωρώ πως χρειάζεται ένα κεντρικό γραφείο ε, διαχείρισης αυτών των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, συντονισμού καλύτερα των επαφών με την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντζέρη. Εγώ παίρνω το λόγο για το νότιο σκέλος ε, της πολιτικής γυτνίασης. Ε, ε, είχαμε θεωρήσει πολλές φορές πολύ σωστή την προσέγγιση του κυρίου Ντέβιντ. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε την κατάσταση διότι στην Μεσόγειο το πλαίσιο όλο ένα και αλλάζει και θα έπρεπε να τονίσουμε ότι χρειάζεται ένα μέσο πολιτικής γυθνίασης πολύ πιο ευέλικτο από αυτό το οποίο έχουμε φανταστεί που θα κρατάει και την αρχή more for more αλλά και θα λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και για να να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τα τρία μη. Money, Market and Mobility. Να μπορούμε δηλαδή να διαπιστώνουμε πάντοτε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ποιες είναι οι προτεραιότητες και όχι να έχουμε απλώς μία ροή βοήθειας ανεξέλεγκτη. Επιμένω, η μεσογειακή πραγματικότητα σήμερα Αύριο δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα μόνο η Τινησία είναι μια χώρα που έχει τους όρους να αλλάξει άμεσα. Χρειάζεται ίσως μια πιο γενναιόδορη πολιτική, σωστά πρικοδοτημένη, ούτως ώστε αυτό το εργαστήριο να μπορέσει να προχωρήσει και να αποτελέσει ένα καλό σημείο αναφοράς για όλη την Αραβική Άνοιξη και να αποφύγουμε σε ορισμένες χώρες αυτή η Άνοιξη να μην καταστεί μεσογειακό φθινόπωρο. Ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Λόκμπιρερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά η κυρία Φλότρεκ, μέρο τη ομάδα μα και ιδιαίτερα για την νότια γειτονία. Ε, ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λιβύη και έτσι δεν μπορεί να μιλήσει. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αναφέρεται μέσα στην έκθεση η κινητικότητα, η διαμόρφωση κινητικότητα ε, στον ε, χώρο τη Μεσογείου και Ιδιαίτερα θα θέλω να επισημάνω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίθηκε η, ανανέωση τη εντολή τη Frontex, πράγμα το οποίο πιστεύω θα πρέπει να μα απασχολήσει. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι είδου πολιτική ε, στα σύνορά μα ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αναπτύξουμε. Επίση θα πρέπει να δούμε τα ιστιτηρότητε των κρατών μελών και τι ανάγκε ε, σε ανάπτυξη του κράτου δικαίου, των δομών, τη δικαιοσύνη ιδιαίτερα. Αυτή είναι οι τρει τομεί που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Ευχαριστούμε την κυρία Λόχ Πίλερ. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ σε αυτήν τη συζήτηση θα συνεισφέρω με ορισμένες τροπολογίες. Αυτή η νέα δυναμική που ανοίγεται σήμερα με ορισμένες χώρες της νότιας όχθης δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Ε, η Μεσόγειος είναι ένας χώρος ε, ασφάλειας. Οι αρχές ε, επανεισδοχής είναι πρώτος στόχος. Όλοι οι μηχανισμοί που έχουμε για τον έλεγχο της μετανάστευσης και για, την, για τους ετούντες στο άσυλο θα πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων αυτών των λαών. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε ορισμένα σημεία, διότι η συνεργασία πάντοτε απευθυνόταν στα κράτη και όλα τα μέτρα ήταν απόλυτα συνδεδεμένα με τα κράτη. Εγώ θα ήθελα να αυξήσουμε την αποκεντρωμένη συνεργασία, κυρίως με την τοπική αυτοδίκηση... διότι αυτή η συνεργασία είχε προβλήματα στο παρελθόν αλλά σήμερα με τις εξωτερικές υπηρεσίες η παρουσία μας είναι πολύ πιο ισχυρή και γίνεται καλύτερος έλεγχος ε, των ε, κονδυλίων. Η αποκεντρωμένη συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των ε, πόλεων, των αστικών περιοχών, των εσωτερικών κοινοτήτων και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σχέδια ζωτικά για τη βελτίωση των όρων ζωής των πολιτών αυτών των χωρών. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τι παρατηρήσει των δύο συναδέλφων από την ομάδα των Πρασίνων. Θα ήθελα να πω κατά βάση ότι όχι μόνο είναι μια καλά διαρθρωμένη έκθεση, αλλά και μια, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορούν ε, να στηρίξουν αυτή την πολιτική γειτονία, τη νέα πολιτική γειτονία, δηλαδή την εταιρική σχέση, τι νέε εταιρικέ σχέσει και όχι μόνο το More for More, αλλά την ανάπτυξη πάνω απ' όλα της ε, κοινωνίας των πολιτών. Και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Σούλτς ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα, μια υπηρεσία, ένα γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο θα διευκολύνει την κοινωνία των πολιτών ε, στις επαφές της και το, και το συντονισμό που χρειάζεται, συντονισμένη εργασία που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν ε, θα έλεγα να μπορεί η κοινωνία των πολιτών να κάνει με την καλή έννοια το λόμπι της καλύτερα. Να μην πρέπει δηλαδή μόνο να περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις δομές της κρατικές ή τις επίσημες των άλλων κρατών. Και επίσης θα ήθελα να προτείνω εκ μέρους των Πρασίνων μια ετήσια αξιολόγηση της ε, ε, κατάστασης των ανθρώπινων δικαιώματα, όχι δυνητικά, αλλά υποχρεωτικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί το could υπάρχει μέσα στο κείμενο ως δυνητικός όρος και δεν υπάρχει το should, θα πρέπει να γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε τη μια χρονιά και όχι την άλλη. Στις ε, διαπραγματεύσεις, στις ε, εμπορικές, αντίθετα με τον κύριο Μιανμό, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε μία μία σύμμετρη σχέση με τις χώρες αυτές, διότι δεν είναι οι συνθήκες αντίστοιχες, οι, τα μεγέθη, οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών, αυτών, δεν είναι συγκρίσιμες. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών αυτών ε, της γειτονίας κατά τρόπον ε, ε, αυτόματο. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Δεν έχω άλλους ε, συναδέλφους εγγεγραμμένους. Υπάρχει κάποιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ήθελε να σχολιάσει. Εάν ναι, θα τον ακούσουμε. Αν όχι, τα τελικά σχόλια στους εισηγητές. Μπροκ και μετά Σίβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις ε, Παρατηρήσεις σχετικέ μεταξύ του κυρίου Ντάβιτ ε, θα τι διαβιβάσω φυσικά. Πιστεύω ότι οι προτάσει που ακούστηκαν σε έναν βαθμό αφορούν και τα δύο τμήματα και τους δύο τομείς. Εν πάση περιπτώσει θα τις διαβιβάσω τις παρατηρήσεις για την πρόταση του κυρίου Σούλτ ε, για το Ίδρυμα. Είναι κάτι το οποίο με απασχόλησε και σε μια συζήτηση που είχαμε τον κύριο Φίλε Ξέρουμε ότι και ο Υπουργό των Εξωτερικών τη Πολωνία ενδιαφέρεται για μια τέτοια εξέλιξη, για ένα τέτοιο ίδρυμα. Θα πάρει όμω κάποιο χρόνο μέχρι να θεσπιστεί. Δηλαδή να σχεδιαστεί, να θεσπιστεί κτλ. Και, και νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι τότε να αξιοποιήσουμε το μέσον για την προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο μα δίνει τη δυνατότητα κατά τρόπο πολύ πιο ευέλικτο να στηρίξουμε τους στόχους αυτούς ε, για την, ε, για την ε, δημοκρατική εξέλιξη, ανάπτυξη, δημοκρατισμό, ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Άπαξ και έχει θεσπιστεί το European Endowment for Democracy, το Ευρωπαϊκό Κατοπίστευμα για τη Δημοκρατία. Νομίζω ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε λίγο πολύ συμφωνήσει σε μια βασική δομή που δεν αφισβητεί κανείς ότι δηλαδή ε, παραδείγματι τα κράτη αυτά της Ανατολικής ε, Γειτονίας ε, πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 49. Αυτό ισχύει και άρα είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει μπορούν να καταθέσουν πρόταση, μάλλον αίτηση στη συνέχεια μετά τις διαπραγματεύσεις. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε συγκεκριμένα τις συμφωνίες συνδέσεις και την εξέλιξη σε χώρους ε, ελεύθερων συναλλαγών, εκεί όπου ενδεχομένως υπάρξει δυνατότητα για περισσότερη συνεργασία, στενότερη συνεργασία και διασύνδεση με κάποια κράτη. Αλλά ας, είναι, ας είμαστε και προσεκτικοί, ας μην δίνουμε ελπίδες, φρούδες και ας μην δημιουργούμε την εντύπωση ορισμένα κράτη ότι μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν. Επίσης, δεν θα πρέπει να δοθεί εντύπωση ότι αυτόματα η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί τον προθάλαμο για την ένταξη ως πλήρους μέλους ενός κράτους. Αυτό θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Δεν πρέπει να ρισμονούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί οι διαπραγματεύσεις να παγώσουν για ένα διάστημα, να σταματήσουν η εξέλιξη αυτή για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις και λύσεις, αλλά δεν θα πρέπει αυτές να γίνουν καθημερινή, ε, καθημερινής χρήσης, να τις προβάλλουμε δηλαδή σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ένα λεπτό κύριε Σίβιτς. Πριν από σας, ο κύριος Νταφ είναι ο εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ και μετά σε εσά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο συγγνώμη που δεν ήρθα νωρίτερα γιατί ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση. Όπως είπατε είμαι ε, συντάκτης νομοδότησης εκ μέρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο βασικά εκείες παρατηρήσεις. Καταρχάς, σε σχέση με την ε, Ένωση για τη Μεσόγειο, είναι απολύτως απαραίτητο να αξιοποιήσουμε σε σχέση με το πλάσμα αυτό, λέει ο μιλητής, ε, όλες τις δυνατότητες που έχουμε διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αυτό το πλάσμα δημιουργήθηκε από κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται τι εστί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν αντιλαμβάνονται τι εστί η Μεσόγειος. Πρόκειται για μία σε θεσμικούς όρους ανομαλία, ανώμαλη κατάσταση και δεν προσφέρει την προσθέμενη αξία που θα απαιτούσε να προσφέρει, θα να προσφέρει μια ευρωπαϊκή πολιτική. Έτσι λοιπόν πρέπει να πω ότι στέκομαι πολύ επικριτικά απέναντι στην ιδέα της συνέχισης της Ένωσης για τη Μεσόγειο στην τωρινή της μορφή. Προτείνουμε δε ή σκοπεύουμε να προτείνουμε Προτείνουμε λοιπόν η ευρωπαϊκή πτυχή της Ένωσης για την ε, Μεσόγειο να υπαχθεί στην αιγίδα ε, στο χώρο αρμοδιοτήτων της κάθε και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μία δεύτερη μεταρρύθμιση που θα θέλαμε να ξεκινήσει μακροπρόθεσμη αυτή τη φορά, μεταρρύθμιση που απαιτεί και αναθεώρηση τη συνθήκης, αλλά αφορά το θέμα του άρθρου 49 συγκεκριμένα, και που αποφεύγουν μάλλον διπλωματικός πως οι δύο συντάκτες της εκθέσεως της ΑΦΕΤ. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι το άρθρο αυτό ενδέχεται η ΑΦΚΟ για μελλοντική αναθεώρηση των, να, να προτείνει μάλλον μια μελλοντική αναθεώρηση της συνθήκης με ιδιαίτερα πρόταση θέσπισης ειδική κατηγορίας μέλους συνδεδεμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αντιστοιχούσε σε τρεις κατηγορίες κρατών κράτη δηλαδή τα οποία δεν δίνανται να ενταχθούν ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν έχουν ε, το χαρακτήρα ευρωπαϊκού κράτους. Δεύτερον, κράτη τα οποία επιλέγουν να μην ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα μπορούσαν ε, τις πράγματι να ενταχθούν. Τρίτον, κράτη τα οποία ενώ προσπάθησαν δεν δίνανται να πληρώσουν τα κριτήρια προσχώρησης. Πιστεύω δε ότι δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε για το μέλλον την συζήτηση θεσμικούς όρους αυτή τη κατάσταση. η πληθώρα σχέσεων αφενός μεν ad hoc, αφετέρου δε εν της πράγμαση de facto ε, που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της επιμένους με ε, άλλα κράτη της γειτονίας δεν μας επιτρέπει πιστεύω να παραγνωρίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αξιόπιστο το πλαίσιο αυτό. Δεν μπορεί να προσφέρει δηλαδή μια μακροπρόθεσμα σταθερή εταιρική σχέση στη γειτονία μας. Αλλά, εν είναι ένα θέμα το οποίο θα υποβάλω για πιο σοβαρή εξέταση στην Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ, κύριε Ντάφ. Ο εισηγητής για το Βορρά, ο κύριος Σίβιτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν, έχει, δεν είναι τελειωμένο το προϊόν αυτό, δεν αποτελεί δηλαδή ολοκληρωμένο κείμενο, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω συζητήσει και βελτίωση και θέλουμε να προσεγγίσουμε όλες τις προτάσεις και ιδέες κατά τρόπον επικοδομητικό. Από τις συζητήσεις που ακούσαμε σήμερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί της ουσίας, μόνο προσπάθεια να βελτιωθεί αυτή η πολιτική έτσι ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τρόπο προγραμματισμένο για το μέλλον. Και θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Όπως γνωρίζετε εσείς και εσείς, τα θέματα τα σχετικά με την προσχώρηση, με τα πλήρη μέλη δηλαδή, καλύπτονται από το άρθρο 14 της εκθέσεως. Πρόκειται για μια διατύπωση που σχετίζεται μετά όσα είπε ο κύριος Μπροκ και χαίρομαι ιδιαίτερως, έτσι συμφωνούμε. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ή Καταπίστευμα για τη Δημοκρατία. Είναι μια νέα ιδέα. Δεν ε, είναι κάτι το ε, παγιωμένο, το δεδομένο. Μια ιδέα που ξεκίνησε μάλιστα από τον Υπουργό των Εξωτερικών της Πολωνίας και βρίσκεται ακόμη στα Σπάργανα. Χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο. Άλλωστε αναφέρεται ξεκάθαρα στο κείμενό μας ότι μπορεί να προσφέρει ε, ε, κάποιο ουσιαστικό κέρδος αυτό το ίδρυμα μόνο εάν συμβάλλει με προσθέμενη αξία στην, στον εκδημοκρατισμό, στα άνθρωπνα δικαιώματα για τις χώρες αυτές. Διαφορετικά δεν έχει κανέναν λόγο ύπαρξης. Εάν η πρικοδότησή του αξιοποιείται ουσιαστικά αποτελεσματικά στοχευμένα και προσφέρει αποτελέσματα, τότε ναι. Εάν όμως μετατραπεί αυτό το ίδρυμα σε ένα γραφειοκρατικό τέρας το οποίο ε, τρέφεται από τις τάχτες του δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν. Για τον κύριο Νταφ και την ανάγκη να προβλεφθεί βάση σύνδεσης ορισμένων κρατών εταίρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε μια περαιτέρω αναθεώρηση της συνθήκης. Είναι μια νέα ιδέα, πρώτη φορά την ακούω, δεν έχω ε, μέχρι στιγμής ακούσει κάτι σχετικό και ως εκ τούτου δεν έχω θέση να εκφέρω αυτή τη στιγμή διότι την έχω μελετήσει αρκετά. Πάντως, εφόσον ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για την ε, καταχώρηση αυτές τις τρεις ομάδες των συνδεδεμένων κρατών που λέτε, των κρατών που θα ε, μείνουν συνδεδεμένα, εκείνα που δεν μπορούν, εκείνα που δεν θέλουν και εκείνα που, που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ε, ίσως να μπούμε σε ένα κυκαιό να αναθεωρήσουν τις συνθήκες. Δηλαδή ε, μπορεί να προσπαθήσουμε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη για να, δώσουμε αυτή, να ορίσουμε αυτή τη νέα κατηγορία συνδεδεμένων μελών, αλλά μην ξεχνάμε ότι εάν κατατάχει ένα κράτος σε μια τέτοια ε, κατηγορία συνδεδεμένου κράτους δηλαδή, δεν θα έχει ευκαιρία να βγει από την κατηγορία αυτή για να γίνει πλήρες Δεν θα προβλέπεται ενδεχομένως κάτι τέτοιο. Και άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιδράσουν τα τρίτα κράτη αυτά ε, και να έχουμε δυσκολίες στο επίπεδο αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο ε, θα συζητήσουμε στις λεπτομέρειές του την έρθει ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σίβιτς. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 7 Οκτωβρίου στις 12. Σημείο 5. Ε, είναι η συνεργασία με την Κεντρική Ασία, ε, το στάδιο της εφαρμογής της στρατηγικής. Ευχαριστώ την κυρία Νίλσεν που δέχθηκε να καθυστερήσουμε το σημείο της. Της δίνω μέσω στο λόγο. Merci, Monsieur le Président. J'ai envie de dire Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω, ήθελα να σας πω ότι αυτή η γνωμοδότηση σε σχέση με το εμπόριο του Βάμβακος στο Ουσμπεκιστάν έχει προχωρήσει. Έχουμε κάνει συσκέψεις με τους σκιώδεις και προχωράμε προς συμβιβαστική λύση. Όπως θα θυμάστε ίσως ο κ. Μπρόκ είχε εκφράσει επιθυμία για συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες της Κεντρικής Ασίας που έγινε, έγινε με τα μέλη των Επιτροπών άφετίπτα και Ντρουά. Ε, Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα και έτσι είχαμε και μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων καθώς και συστάσεις ε, που μας βοήθησαν να συντάξουμε την έκθεση. Είμαστε στην ίδια γραμμή με την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξη για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Κιλνίλσεν και τώρα έχω τη χαρά να σας δώσω το λόγο με, τον, ε, με την κυρία ε, Γέγκλε, στην κυρία Γέγκλε που είναι σκιώδη ε, συγγήτρια για το ΕΛΚ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Κιλίλσεν για την έκθεσή της. Ήταν καλή, πολύ καλή η συνεργασία μαζί της συνεργασία που είχε σε γνώμονα το στόχο μας για μια καλή έκθεση έντελ. Η κυρία Κιλνίλσον αλλά και εμείς καταθέσαμε τροπολογίες 192 συνολικά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά, δηλαδή να συνδυάσουμε τις προτάσεις περιλαμβάνοντας τις τροπολογίες ε, και να καταλήξουμε σε ένα καλό σύνολο με την έκθεση τελική της μορφή. Πιστεύω, ωστόσο, ότι η ευρύτερη πλειοψηφία των μελών μας θα υποστηρίζει τις ε, τροπολογίες αυτές. Με συγχωρείτε. Πρόεδρε, μιλάμε για τη γνωμοδότηση για τον βάμβακα του Ουσμπεκιστάν ή την έκθεση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία. Τα μπέρδεψα. Εγώ άρχισα να μιλάω για τη γνωμοδότηση σχετική με το Βάμβακα και όχι για την ε, Κεντρική Ασία. Το 5 μιλάει για την στρατηγική για την ε, Κεντρική Ασία. Γι' αυτό μιλάμε κανονικά. Μάλιστα, έκθεση. Και όχι για τη γνωμοδότηση, όχι για το βαμβάκι. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Σύμφωνοι. Ναι, για την έκθεση μιλάμε, κύριε Γέγκ. Πρόεδρε, αν μιλάμε για την έκθεση, προτείνω και πάλι να λάβει το λόγο η κυρία Κιλνίλσεν, αφού είναι η συγγήτρια. Μάλιστα. Έκθεση. Για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία. Λέει η κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, την κυρία Γέγκλε, ιδιαίτερος, που έλαβε ενεργό μέρος στη δουλειά αυτή. Οι προτάσει αυτέ που μα έκανε ενισχύουν το κείμενό μα. Είχαμε προτάσει και από τον κύριο Σπαβόντα, την κυρία Κοπά και άλλου συναδέλφου που μα έστειλαν τι προτάσει του. Αυτό δεν θα ήθελα να πω εγώ σήμερα. Είναι ότι στην έκθεση αυτή, στη φάση της σύνταξης του κειμένου, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τη δομή που είχε η προηγούμενη έκθεση για τη στρατηγική ε, της σε σχέση με την Κεντρική Ασία του 2007 την έκθεση δηλαδή όχι για λόγους ευκολία, αλλά γιατί θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση αυτή να δούμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση με, ε, σε σχέση με διάφορα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Το μήνυμα λοιπόν που ακούσαμε τόσο εκ μέρου των επισήμων εκπροσώπων των διαφόρων χωρών αλλά και των διαφόρων ενώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν αυτή η ανάγκη του να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας, τη βοήθειά μας, τη συνεργασία ανάλογα με τον βαθμό ανοίγματο της κάθε χώρας Θεωρήσαμε λοιπόν σημαντικό να στείλουμε ειδικέ παρατηρήσεις στην Υπηρεσία Εξωτερικών, ειδικά για την κάθε χώρα. Και επιμένω σε αυτό το σημείο, διότι υπάρχουν μερικά μικροπροβλήματα με ορισμένου συναδέλφους και θέλω τα πράγματα να είναι σαφή. Αυτό λοιπόν το τμήμα της έκθεσης που προχωρεί σε μία διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω σήμερα επέμεινα για, γύρω από το θέμα της ασφάλειας αλλά η ο όρος ασφάλεια στην Κεντρική Ασία ε, ερμηνεύεται ως ασφάλεια του υπάρχοντος καθεστώτος εμείς εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη ασφάλεια, για την προώθηση της ασφάλειας υπέρ του πληθυσμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση. Στο επίκεντρο των προγραμμάτων μας θα πρέπει να έχουμε αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή. Θα δώσει μεγαλύτερη νομιμότητα και ευστοχή αποτελεσματικότητα στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Όλοι οι συνάδελφοι συμφωνήσαμε 100% γύρω από αυτά τα δύο σημεία της έκθεσης. Νομίζω ότι η κυρία Γέγλερ μπορεί να πει μερικά πράγματα γύρω από αυτά, αλλά ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα προταθεί μία συνεδρίαση για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γέγελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν είναι βέβαια εύκολο να ε, δούμε τα θέματα χωριστά το ένα από το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ καταρχάς την κυρία Κιλ Νίλσεν. Όλες αυτές οι τροπολογίες, όπως είπε, μας υποχρεώνουν να τηρήσουμε μια γραμμή ενιαία και συνεκτική. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικέ μέσα από τι τροπολογίε αυτέ και βελτιώνουν σημαντικά το κείμενο και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε χάρη στην καλή μα συνεργασία να καταλήξουμε σε ένα ε, πολύ καλό κείμενο. Οι σχέσει λοιπόν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Ασία ε, προβάλλονται σε πολλέ από τι τροπολογίε και αυτό είναι και ένα αίτημα, ε, ένα ζήτημα που θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ιδιαίτερω η Κεντρική Ασία είναι ένας χώρος μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και όλα αυτά τα κράτη της Κεντρικής Ασίας στρέφουν το βλέμμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτούν εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο τα κράτη αλλά και οι άνθρωποι οι ίδιοι, τι κάνει και πώς στέκεται και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να τους ε, να, να ανταποκριθούμε και εμείς. Ιδιαίτερα λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδιαίτερα όλες αυτές οι έννοιες που υπάγονται στον τίτλο «Εκδημοκρατισμός» είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Πολλές είναι οι εξελίξεις ωστόσο που μας οδηγούν στο συμπεράσμα ότι χωρίς καλή οικονομική εξέλιξη δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν και συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες ασφαλείας για τους πολίτες ικανοποιητικές. Και γι' αυτό ο εκδημοκρατισμός μαζί με την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να εξετάζονται. Δεν μπορούν δηλαδή να αποκοπούν η μία έννοια από την άλλη. Η ε, διαφοροποίηση επίσης των οικονομικών σχέσεων έχει πάρα πολύ σημασία. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε μόνο ή να δώσουμε την εντύπωση ότι ασχολούμαστε μόνο με, τους, ε, με το φυσικό πλούτο σε πρώτες ύλε των κρατών αυτών. Πρέπει να στηρίξουμε και την ανάπτυξη παραγωγικών ε, μονάδων και διαδικασιών στις αυτές τις χώρες για τα επιμέρους κράτη. Τουρκμενιστάν, Καζαχστάν. Γίνονται επιμέρους ε, παρατηρήσεις. Εδώ θα ήθελα να πω εν γέννη για όλα τα κράτη της Κεντρικής ε, Ασίας ότι ε, πρέπει να συνομιλούμε μαζί τους ως ίσως προς ίσον και ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να, την, τον πειρασμό ή την τάση να επιβάλλουμε ε, στοιχεία του δικού μας πολιτισμού και της δικής μας κουλτούρας, ή νοοτροπίες στα κράτη αυτά, αλλά να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν και να αναπτυχθούν μόνα τους. Κάποιες λοιπόν προτάσεις μπορούν να συμπληρωθούν ε, με τις τροπολογίες. Θα καλέσουμε βεβαίως τις κυβερνήσεις ε, να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ζήτημα και της μετανάστευσης αλλά και της διαχείρισης των φυσικών πόρων, υδάτων κτλ. και ιδιαίτερα θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη βούληση, την ε, έκκληση για μια σαφέστερη βούληση για μεταρρυθμίσεις. Οι δε πρεσβείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχετικά κράτη στα κράτη της Ασίας, της Ασίας δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο ως προτάσεις επί χάρτου, αλλά να υλοποιηθούν και να επανδρωθούν ε, και να εξοπλιστούν κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις που συνεπάγεται η ανάληψη των δραστηριοτήτων τους. Ε, Επίση, θα έπρεπε, πιστεύω, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις μεταξύ βουλευτών και σε ισότιμους όρους για την προαγωγή και των σχέσεων φιλίας αλλά και σεβασμού μεταξύ ημών και των κρατών αυτών. Όπως είπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Συνεχίζεται ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από τη δική μου προσωπική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια μπορώ να δηλώσω ξεκάθαρα ότι υπάρχει σαφής πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα παρότι παραμένουν αρκετά προβλήματα ακόμη σε όλα αυτά τα κράτη. Η κυρία Κιλνίσελ ε, είχε προχτές ε, συζήτηση με εκπροσώπους της UNICEF για το θέμα μεταξύ άλλων της παιδικής εργασίας και την οποία τη θεώρησε πάρα πολύ χρήσιμη για την έκθεση αυτή. Θέλουμε να αναπτύξουμε προγράμματα στον τομέα της ανάπτυξης που θα σημαίνουν επενδύσεις, που σημαίνουν περισσότερη υποστήριξη για την διαβίου μάθηση Φερρυπίν και αφενός αλλά και ε, υποστήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης για παιδιά αλλά και νέους, κυρίως στον χώρο της υπαίθρου και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές αφετέρου. Όπως είπε η κυρία Κιλ Νίλσεν, ε, συνεχίζουμε τη συνεργασία. Έχω ακόμα μία πρόταση που δεν είχα διατυπώσει. Τώρα μόλις άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει αυτή η ιδέα στο μυαλό μου το TIEX, το Twinning και το Sigma μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν έχουν ακόμη επεκταθεί στα κράτη, στη σχέση με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας αλλά που στηρίζονται, ε, στηρίζουν μάλλον ε, κράτη ε, με συμφωνίε συνδέσεις ή υποψήφια για ένταξη στην ε, πρόοδό τους. Ίσως θα έπρεπε αυτά να τα δούμε σαν προτάσεις ε, για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτα κράτη. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω προφορικώς να καταθέσουμε τη σχετική τροπολογία και να επιτρέψουμε την ανάπτυξη ενός πεδίου αναλογισμού για την ε, πρόταση αυτή. Ίσως θα μπορούσαμε να ε, ρωτήσουμε και τις απόψεις των ενδιαφερομένων ε, για, το, για τις προτάσεις αυτές, να τις σχολιάσουν. Ευχαριστώ κυρία Γέγελ. Δεν, θέλω να μιλήσει, θέλει να μιλήσει η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυρία Κιλνίσε για τα τελικά σχόλια. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Διαπιστώνω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος ε, γύρω από αυτή την έκθεση η κυρία Γιάγελ έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μία πρόταση για αυτό το κοινοβουλευτικό περιφερειακό φόρουμ το οποίο θέλουμε να προτείνουμε στις χώρες της Κεντρικής Ασίας που θα επιτρέψει ταυτόχρονα ανταλλαγές μεταξύ βουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά και των βουλευτών της Κεντρικής Ασίας θα μπορέσουν να, διαλο... να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους οι βουλ... κεντρασιάτες βουλευτές για δικά τους περιφερειακά προβλήματα. Η τελευταία πρόταση ε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον με πλήσετε με τη νέα σας πρόταση, δεν θα σας απαντήσω τώρα, φυσικά και θα το συζητήσουμε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη όταν διαπιστώνω ότι η κοινή λογική που διέπει τις εργασίες μας είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κιλ Θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα στην γνωμοδότηση, πάντα είναι η συγγήτρια η κυρία Κιλνίτσεν σχετικά με την επέκταση των διατάξεων της συμφωνικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ουζουμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο, διμερές εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά στο κλώστο υφαντουργικό εμπόριο το συζητάει και η Ίντα και η, και η ε, Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, παιδική εργασία ε, στα χωράφια καλλιέργειας βαμβακιού εργάζονται τα παιδιά. Εμείς το συζητάμε, ναι, εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά συνεδριάσαμε από κοινού και με την Ίντα και με την Τρόη με εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν διευκρινήσεις και συστάσεις, συγκεκριμένες συστάσεις για να μειώσουμε, να περιορίσουμε αυτή την πρακτική της καταναγκαστικής εργασίας των παιδιών στο Ζουμπεκιστάν. Και εδώ φαντάζομαι θα καταλήξουμε σύντομα σε έναν συμβιβασμό. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις από τους συναδέλφους. Α, κυρία Βεβαίω. Έχετε το λόγο κυρία Γιώργη. Συγγνώμη πρόεδρε. Και τώρα εκφράζω την κυρία Βάιντερε και εκπρόσωπό που είναι η σκιώδη η συγγετριά μας δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Για την έκθεση αυτή λοιπόν και πάλι ευχαριστώ την κυρία Κιλνίλσεν πρόκειται για μια έκθεση που ε, αφορά κυρίως την ίντα βέβαια είναι επί της ουσίας αρμόδια ίντα. Ωστόσο ήθελα να πω ότι χωρίς να έχουμε ριζικά αντιθέτες θέσεις διαφοροποιούμαστε. Για το ΕΛΚ δεν έχει νόημα ε, να τεθούν φραγμοί στην λειτουργία αυτής της συμφωνίας και να ε, πούμε ότι θα πρέπει πρώτα να σταματήσει η εκμετάλλευση παιδικής εργασίας ε, και να πάψουν όλα τα άλλα προβλήματα και μετά θα αναπτύξουμε τις εμπορικές σχέσεις. Το Σμπικιστάν τους άλλους εμάς δεν μας χρειάζεται για το εμπόριό του, έχει την Κίνα έχει το μπαμπάκι του να πουλήσει και θα το πουλήσει όπως και να έχει. Ε, θα ήθελα λοιπόν μαζί με τους άλλους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού ε, Λαϊκού Κόμματος να σημειώσω ότι και αυτό ισχύει βέβαια όχι μόνο για το Ουσμπικιστάν αλλά και για το Τουρκμενιστάν σε άλλες ε, σχέσεις και με άλλα κράτη ότι θα πρέπει χωρίς να παγώσουμε ή να διακόψουμε τις εμπορικές σχέσεις να συνεχίσουμε την συνεργασία και τις προσπάθειες. Γιατί από τους ε, εκπροσώπους της UNESCO με χαρά άκουσα προχτές ότι έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Ουσμπεκιστάν, ότι κάνουν τα σχόλιά τους, ε, ότι επικρίνουν βεβαίως ε, την παιδική εργασία και την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, αλλά από την άλλη έχουν πέσει τα νούμερα χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικά, γιατί από τα 2 εκατομμύρια έχουν πέσει το 1 εκατομμύριο τα παιδιά που δουλεύουν. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, τότε μπορούμε να πούμε ότι με αυτέ τι εμπορικέ σχέσει θα έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα για του ανθρώπου τη χώρα αυτή, που σε τελευταία ανάλυση μπορούν να τα επενδύσουν μετά για να αγοράσουν οι μηχανέ και έτσι να μην χρειάζεται πια η παιδική εργασία. Δηλαδή μπορεί και αυτό ακόμη να βοηθήσει σε μια θετική εξέλιξη και ένα σημείο το οποίο θα ήθελα εξάπαντος να απορρίψω σαν πρόταση, σαν διατύπωση, είναι η έννοια που αναφέρεται στο κείμενο η χειρότερη δικτατορία του κόσμου. Μπορεί κανεί να έχει την άποψη αυτή για το Ουσβέκισταν, αλλά το να λέμε ότι μια χώρα είναι η χειρότερη δικτατορία του κόσμου σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω δεν έχει θέση. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τα άλλα όμω νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Κιλίνη. Ευχαριστώ κυρία Γιάγκελ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Κύριο Σίβιτς. Κύριε Σίβιτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αντικαθιστώ την Ελένη Κοπά. Λόγω των αλλαγών στην ημερήσια διάταξη δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την θέση της ομάδας μας αυτοπροσώπως και την αντικαθιστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ενώ συμμεριζόμαστε τις επικρίσεις για τις λύσεις που εφαρμόζονται από την ε, κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν σε σχέση με τους παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, θα ήθελα ιδιαίτερως να τονίσω ότι υπάρχουν αποδεδειγμένες περιπτώσεις όπου παιδιά χρησιμοποιούνται και είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας και αυτό αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο. Γι' αυτό αυτό που θα ζητήσουμε είναι οι αρχές της χώρας να σταματήσουν οριστικά την εκμετάλλευση των παιδιών. Εμείς ως σοσιαλιστές θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Σίβιτς. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος ε, της εξωτερικής υπηρεσίας που θέλει το λόγο. Ούδης. Ωραία. Ψηφίζουμε στις 4 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Μπορούμε λοιπόν να αποχαιρετιστούμε. Ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση 4 Οκτωβρίου στις 3. Σας ευχαριστώ. Καλή επάνωδο.